Έχουμε διερμηνείς που να δουλεύουν σε όλες τις γλώσσες. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το συμβάν. Δεν ξέρουμε ακριβώς από τι προκλήθηκε. Σε κάθε περίπτωση δεν ήμασταν καθόλου σε κίνδυνο. Και ε, εκτιμώ ιδιαίτερο το γεγονός ότι όλοι ε, συνεργάστηκαν και εγκατέλειψαν την αίθουσα της Ολομέλειας για λόγους ασφαλείας και ε, άφησαν το χώρο ελεύθερο για να τον ελέγξουν οι υπηρεσίες ασφαλείας. Και αυτή την ενημέρωση έχω από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Προεδρείου.